Καλημέρα σας. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τις απογευματινές μας εργασίες, γιατί τελικά αν δεν ξεκινήσουμε, έστω και αργοπορημένα, δεν θα μπορέσουμε να σεβαστούμε όλο το, όλο το πρόγραμμά μας. Πρώτο σημείο λοιπόν στην ημερήσια διάταξη της απογευματινής συνεδρίας Είναι μια δικιά, μας, δικιά μου ε, έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με την συνέχεια που πρέπει να δοθεί στην ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και τον έλεγχο των το κράτη-μέλη της άσκησης εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή. Στην ουσία μάλλον είναι γνωμοδότηση. Η εισηγητής ε, είναι στην αρμόδια επιτροπή, στη Γιούρη δηλαδή, ο συνάδελφος Γιώζεφ ε, Σάγερ. Και η δικιά μας επιτροπή, μαζί με πολλές άλλες, ε, πρέπει να εκπονήσει γνωμοδότηση σχετικά με το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων και των κατεξουσιοδότηση πράξεων κτλ. Μου έκανε την τιμή η επιτροπή μας να με ορίσει εισηγήτρια. Σε αυτήν την ε, πρώτη μου γνωμοδότηση και με τη βοήθεια βεβαίως της ε, ε, γραμματείας αποφάσισα να περιορίσω το εύρος της γνωμοδότησης, δηλαδή να ασχοληθώ με τον τρόπο με τον οποίο μέχρι τώρα η Επιτροπή δική μας αντιμετώπισε το ζήτημα αυτό. βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι ρυθμισμένο ακόμα το κεφάλαιο αυτό και επομένως προκύπτει ανάγκη να βρούμε μία ενιαία αντιμετώπιση του ζητήματος από τις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Για τις τροπολογίες να σας πω ότι η 2 Ιουλίου του 2013 στις 12 το μεσημέρι είναι η προθεσμία. Ε, για την υποβολή τροπολογιών. Ψήφο στην Επιτροπή μας 18 Σεπτεμβρίου, ψήφο στην Ολομέλεια ε, Νοέμβριο του 2013. Ε, πρόκειται για ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά εάν κάποιος θέλει να μιλήσει, παρακαλώ, έχει το λόγο, όποιος επιθυμεί, διαφορετικά μπορεί να εκφράσει την άποψή του μέσω της υποβολής τροπολογιών. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν πολλά σχόλια. Σας προτείνω λοιπόν να διαβάσετε αυτήν την εργασία. Ε, δεν μπορώ να την παρουσιάσω γιατί είμαι και πρόεδρος ε, σήμερα. Διαβάστε λοιπόν τις προτάσεις που κάνω ε, και μετά θα δούμε ποια είναι, ποιες είναι οι τροπολογίες τις οποίες θα υποβάλουν και ποιο θα είναι το πνεύμα τους, ποιες τροπολογίες θα υποβάλουν οι συνάδελφοι. Ναι, παρακαλώ. Πολύ γρήγορο σχόλιο θέλω να κάνω. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τις ε, ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις, αλλά να μην ε, λησμονήσουμε, να δούμε και την αναλογικότητα. Πόσες είναι μία, δεκαπέντε, δεκαέξι. τότε αν είναι έτσι μπορεί χωρίς συναπόφαση να, να προχωρήσει όλη η νομοθεσία, όλο το νομοθετικό έργο. Επομένως θα πρέπει να δούμε ποια είναι η αναλογικότητα έτσι ώστε να μην χάσουμε τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες που έχουμε σαν κοινοβούλιο. Επομένως όχι μονάχα ε, να δούμε ε, τι είδους είναι η κατεξουσιοδότηση πράξης αλλά και πόσες, ποια είναι η αναλογία τους. Γιατί αν έχουμε 16 ας πούμε κατά εξουσιοδότηση πράξη μια ε, οδηγία, δεν λέω ότι είναι ούτε πολλά ούτε λίγα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει ο λόγος, η, η, η σχέση να είναι σωστή και αναλογική. Και νομίζω ότι αυτό το σημείο μπορείτε λίγο να το εμβαθύνετε. Ευχαριστώ. Φυσικά λέει η Πρόεδρος, φυσικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί σκόπιμο να πάρει το λόγο επί του θέματος αυτού. Θέλει να μας πει κάτι. Από ό,τι φαίνεται όχι. Λοιπόν, ε, να παρακαλέσω τους συναδέλφους να διαβάσουν αυτό το προσχέδιο το οποίο έχω προετοιμάσει και να ε, σκεφτούμε επίσης ε, και να σκεφτούν οι συνάδελφοι ότι μέχρι τις 2 Ιουλίου έχουν περιθώριο για να υποβάλουν τις τροπολογίες τους. Allora, oggi sembra una giornata Είναι δύσκολη η μέρα σήμερα. Δύσκολη η μέρα, τι να σας πω. Έχουμε το επόμενο σημείο για το οποίο η συγγήτρια είναι η κυρία Νίμπλερ η οποία μόλις μας ειδοποίησε ότι θα φτάσει με ελαφρά αργοπορία. Πέντε λεπτάκια. Επομένως θα ε, σταματήσουμε για πέντε λεπτά. Είναι μια καλή ώρα για να πεταχτείτε να κάνετε κάποιο τηλεφώνημα αν θέλετε ή κάτι τέτοιο ναι. λέει η πρόεδρος. Και μόνο ακόμα ένα σημείο μετά την κυρία Νίμπλερ έχουμε ακόμα ένα σημείο από ό,τι φαίνεται. Α, όχι, δύο, δύο. Εντάξει. Σε του.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 Λοιπόν, να αρχίσουμε με το σημείο 10 και να δώσω μέσα το λόγο στη συνάδελφο Χέρτσκοκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είσαστε εσείς εδώ, ο σκιώδης μου συγητής επίσης και όλοι αυτοί οι οποίοι είναι παρόντες ε, βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή Πολλοί άλλοι ενδιαφερόμενοι είναι στην Επιτροπή, προσωπικού, στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Θα ήθελα να κάνω μια εισαγωγική παρέμβαση για το πώς βλέπουμε το κεφάλαιο 108 στο πλαίσιο αυτό. Και να σας πληροφορήσω για την αίτηση του κυρίου Λαμασούρ προς την Επιτροπή μας να διατυπώσουμε μια επιστολή όπου θα οριστικοποιήσουμε τις σκέψεις μας για το κεφάλαιο 1α, συγγνώμη, όχι 108. Φαίνεται ότι κοντεύει να κλείσει πια αυτό το κεφάλαιο και παρά το γεγονός ότι δεν μας ικανοποιούν τα αριθμητικά στοιχεία, δεν θα είμαστε σε θέση να διαφυσβητήσουμε τα συγκεκριμένα αυτά ποσά. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε στα πλαίσια της γνωμοδότησής μας προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών είναι το θέμα της προστασίας των σχεδίων που θέλουμε να διατηρήσουμε τη χρηματοδότησή τους με τη μέθοδο του ring fencing και η επιστολή που έχουμε προετοιμάσει αναφέρει ότι πρέπει να προστατευτεί το ίτερ ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί το υπόλοιπο, το υπόλοιπο τμήμα του κεφαλαίου 1α ή τα, τα περιθώρια μέχρι τις οροφές των δημοσιονομικών προοπτικών για να χρηματοδοτήσουν το ίτερ. Εμείς βέβαια δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τη χρήση των περιθωρίων, αλλά μπορούμε στην επιστολή που θα στείλουμε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών να αναφέρουμε ότι έχουμε προτεραιότητες για την χρήση των περιθωρίων μέχρι τις οροφές στην κατηγορία αυτή και η πρότασή μου είναι να χρησιμοποιηθούν μονάχα για σχέδια τα οποία προωθούν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και για να δώσουμε έμφαση στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για θέματα έρευνας. Με άλλα λόγια, δεν νομίζω δεν νομίζουμε ότι τα υπόλοιπα χρήματα από την ε, για το Connecting Europe Facility θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το περιθώριο αυτό. Κατά τα άλλα πιστεύω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε ως Επιτροπή Ήτρε ότι εάν δεν υπάρχουν οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις για το κεφάλαιο 1α θα πρέπει να ζητήσουμε από την Κομισιόν να μας παρουσιάσει ιδέες για το πώς το κανονιστικό πλαίσιο μπορεί να τροποποιηθεί για να είναι πιο αποτελεσματικό και να παροτρύνουμε την Κομισιό να μας παρουσιάσει προτάσεις σε διαφόρους τομείς που έχουν να κάνουν με τη βιομηχανική πολιτική, την ενεργειακή πολιτική, την πολιτική τηλεπικοινωνιών και τα λοιπά. Ώστε να εξοικονομήσουμε κάποια ποσά. Και τέλος, νομίζω θα πρέπει να υπενθυμίσω για τις επενδύσεις στην κοινωνία της γνώσης και του επιχειρήν ότι είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε αυτές τις ε, επενδύσεις. Προφανώς δεν έχουμε νομικό δικαίωμα να προστατεύσουμε τα περιθώρια, αλλά θα έπρεπε να αναφέρουμε ποιες είναι οι προτιμήσεις μας για να αντιμετωπίσουμε την περικοπή του προϋπολογισμού που έχει προέλθει. Αυτά ήθελα να πω. Και αν συμφωνείτε, νομίζω ότι αυτή η επιστολή μπορεί να σταλεί από την πρόεδρο όμως την κυρία Σαρτόρη, η οποία θα το υπογράψει και θα το στείλει το ταχύτερο δυνατό στον κύριο Λαμασούρ. Er. Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε Ερτσκοκ. Θέλει κάποιος συνάδελφος να προσθέσει κάτι, να σχολιάσει, όχι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως κάποιος εκπρόσωπός της είναι παρούσα. Ναι, είναι παρούσα. Δεν θέλει όμως να παρέμβει, άψογα. Επομένως, μια και κανείς ε, δεν ε, ε, θέλει να παρέμβει περαιτέρω και αν συμφωνεί και η συνάδελφος Χέρτσκοκ να στείλουμε όπως ετήθηκε η ενδιαφερόμενη αυτή την επιστολή στον πρόεδρο Λαμασούρ. Ωραία λοιπόν. Τερμινάτο. Ολοκληρώθηκε και η εξέτωση του σημείου 10 της ημερησίας διατάξεως και επομένως αναμένουμε την συνάδελφο Αγγέλικα Νίμπλερ. Και l'ultimo punto all'ordine del giorno. On attend Ωραία, φτάσαμε στο σημείο 9 της ημερησίας διατάξεως. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Νίμπλερ, στην οποία δίνω αμέσως το λόγο. Και το θέμα της είναι η διαστημική βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ κυρία Νίμπλερ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη φυσικά από τους συναδέλφους γιατί καθυστέρησα, γιατί ήμουν σε μια άλλη επιτροπή και δεν ήθελα όμως να σας καθυστερήσω. Συμφωνήσαμε ότι σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν για τη Διαστημική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συντάξουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας και χαίρομαι που έχουμε και πάλι την ευκαιρία σήμερα να έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψε ώστε να μπορέσω να πάρω και τις προτάσεις και τις ιδέες των συναδέλφων που είναι παρόντες. Να ήθελα, θα ήθελα να πω καταρχήν το εξής, ότι εγώ χαιρετίζω ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Κομισιόν έχει υποβάλει αυτήν την ανακοίνωση για την διαστημική βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τύχει την της αντίστοιχης σημασίας και είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Η βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να ασχοληθεί ιδιαίτερα για το διάστημα. Σε επίπεδο περιεχομένου, να σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση, η πολιτική διαστήματος, όπως ξέρουν πολλοί συνάδελφοι, έχει πάρει ένα πολύ πολύ πλοκό χαρακτήρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καταρχήν γιατί υπάρχουν πολλοί εμπλεκόμενοι, στην αγορά των προϊόντων αυτών. Δεν έχουμε μια κλασικού χαρακτήρα αγορά. Καταρχήν έχουμε στην Ευρώπη ένα αριθμό επιχειρήσεων που μπορούν να ανταγωνιστούν σε κάποιο βαθμό τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου η διαστημική βιομηχανία είναι στρατιωτικού χαρακτήρα κυρίως και είναι πολύ δύσκολο να καθορίσουμε σε τι ακριβώς συνίσταται η διαστημική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει πέντε συγκεκριμένους στόχους για αυτή τη βιομηχανία. Καταρχήν να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό και σταθεροκανονιστικό πλαίσιο. Δεύτερον, να υπάρξει μια ανταγωνιστική, αποτελεσματική και στεναρή βιομηχανική βάση της Ευρώπης, η οποία θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τρίτον, να εξασφαλίσουμε το συγκεκριμένο στόχο της παγκόσμιας αναγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής διαστημικής βιομηχανίας, ώστε να γίνει το μέσο αυτός πιο αποδοτικός οικονομικά σε ό,τι αφορά την παροχή προσθέμενης αξίας, επίσης την να αναπτύξουμε αγορές για δορυφορικές υπηρεσίες και εφαρμογές και τέλος, αλλά όχι ο ιστατός στόχος, το να εξασφαλίσουμε μια τεχνολογική ανεξαρτησία και την ανεξαρτησία σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των ευρωπαϊκών φορέων στο διάστημα. Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, η Κομισιόν έχει προτείνει μια σειρά από μέτρα. Δεν χρειάζεται τώρα να σας αναφέρω όλα αυτά τα μέτρα, γιατί μπορείτε να διαβάσετε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολιτικά όμως θέλω να πω ότι για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι από αυτούς τους 37 τομείς ε, δράσεως θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια σειρά προτεραιοτήτων. Να δούμε ποιο είναι το πιο σημαντικό, πού εμείς θα πρέπει να θέσουμε την έμφαση, πού έχουμε εξάλλου και τη δυνατότητα εμείς ως Ευρωπαίοι να παίξουμε και κάποιο ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο. Παραδείγματος χάρη τι ρόλο παίζει η ευρωπαϊκή πολιτική για το φάσμα των συγνωτήτων σε ό,τι αφορά τη διαστημική πολιτική και ποιε θα πρέπει να είναι οι ερευνητικέ μας δραστηριότητε που συνάπτονται με το ορίζον 2020, πώς να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτές τις δραστηριότητε για να συμβάλλει στους στόχους του 2020, τι ρόλο πρέπει να παίξουν φόρεις όπω η ΕΣΑ, τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, <clears throat> πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών φορέων και των εθνικών κρατών. Λοιπόν, πρόκειται για μία πλειάδα θεμάτων και προβλημάτων από, για, όλα αυτά τα ερωτήματα πρέπει να δώσουμε μία πολιτική απάντηση και φυσικά εγώ περιμένω να ακούσω και τις απόψεις όλων των συναδέλφων που θα μας βοηθήσουν να καταλήξουμε σε ένα οδικό χάρτη βάσει του οποίου θα μπορέσουμε να κατευθύνουμε και την βιομηχανίας, τις κέρυες επενδύσεις που απαιτούνται σε αυτό το νευραλικό τομέα και θα εξασφαλίσουμε και κάποια σταθερότητα και ασφάλεια για το σχεδιασμό. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας θα πρέπει να δώσουν μια ε, συμβολή για το θέμα αυτό. Στο τέλος, σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, εγώ θα προσπαθήσω να δώσω την έκθεση μου στη μετάφραση στις αρχές του Αυγούστου, ώστε να είναι διαθέσιμη στις αρχές Σεπτεμβρίου και εάν συμφωνείτε προτείνω να τεθεί η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες στις 4 Σεπτεμβρίου ώστε στις 26 Σεπτεμβρίου να μπορέσουμε να ψηφίσουμε την έκθεση αυτή και μετά να περάσουμε στην Ολομέλεια ώστε ήδη εφέτος να μπορέσουμε να περάσουμε αυτό το θέμα στην Ολομέλεια <clears throat> και να έχουμε τη δυνατότητα επομένω να έχουμε κάποια επιρροή στην περαιτέρω εξέλιξη αυτής της πολιτικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την ε, συνάδελφο Νίμπλερ. Το λόγο έχει ο ε, συζητητής κ. Ρέμικ. Ευχαριστώ. Θα ήταν κρίμα να μην ε, σχολιάσω αυτό το θέμα. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ μαζί σας λοιπόν και χαίρομαι που υπάρχει για ένα τέτοιο κείμενο επιτάπητος. Είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι η εισηγήτρια ήταν το κατάλληλο άτομο να αναλάβει αυτή την έκθεση. Η κυρία Νίμπλερ τα γνωρίζει αυτά τα θέματα. Είμαι σίγουρος ότι τα αποτελέσματα θα είναι εξαιρετικά. Αυτή η έκθεση θα μας δώσει τη δυνατότητα να αναλύσουμε πολλά προβλήματα και να συγκεντρώσουμε τις σκέψεις μας και σε ένα βαθμό να συμφωνήσουμε επί των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσουμε θεωρώ ότι είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ε, τομείς ε, και μέσα από τη διάθεσή της Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρήσουμε τον ηγετικό μας ε, ρόλο, τον οποίο έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες γιατί δεν είχα τη δυνατότητα να μελετήσω τα κείμενα της Επιτροπής σε βάθος. ασχολούμαι με αυτά τα ζητήματα από τότε που ήρθα σε αυτό το κοινοβούλιο και ήδη βρίσκομαι στη δεύτερη μου θητεία. Πάντα λέω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε την πρόσβαση στο διάστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μελλοντικές γενναίες. Γιατί ε, αυτό θα αποτελέσει απαρχή για πολλά άλλα ζητήματα. Πρέπει να δούμε και τι κάνουν οι υπόλοιποι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΗΠΑ και Ρωσία ουσιαστικά. Οι μεγάλες δυνάμεις που είναι σε θέση να εκτοξεύουν αντικείμενα στο διάστημα. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Θα σταματήσω εδώ και βεβαίως προσβλέπω σε συνεργασία με την εισηγήτρια και είμαι διατεθειμένος να συμβάλλω στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Στην ψηφοφορία στις 26 Σεπτεμβρίου σίγουρα θα είναι ένα πολύ καλό δώρο γενεθλίων για μένα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Πρόντι έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και την συνάδελφο Νίμπλερ ε, καθώς επίσης και τον συνάδελφο Βέρεκ Εγώ διάβασα πολύ γρήγορα, το, έτσι πρόχειρα, το έγγραφο της Κομισιόν. Παρ' όλα αυτά δεν θεωρώ ότι έχει υπάρξει ιδέουσα προσοχή για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι διαστημικές μας ε, υποδομές. Αναφέρομαι ε, ιδιαίτερα στο θέμα των διαστημικών... Ε, La probabilità di collisione E των, διαστημικών αποβλήτων. Ε, αυτή τη στιγμή πρέπει να πω ότι μεγαλώνει όλο και περισσότερο η εξάρτηση που έχουμε από το διάστημα και επομένως ε, πρέπει να αναρωτηθούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε την ασφάλεια των δορυφόρων μας. Γιατί οι απειλές είναι πολλές και σοβαρές. Γίνονται όλο και πιο πιθανές αυτές οι απειλές. Ε, γίνονται διάφορες ε, συγκρούσεις ε, και σε κάθε σύγκρουση τα απόβλητα όπως και τα αποκολόμενα τμήματα είναι πολύ μεγάλα. Και βλέπουμε ότι αυτές οι περιπτώσεις αυξάνονται με γεωμετρικό ρυθμό. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό και μάλιστα θα έλεγα να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε τώρα. Να αρχίσουμε ε, να ε, ξεκινήσουμε από τώρα δηλαδή ε, μία προσπάθεια καθαρίσματος του διαστήματος έτσι ώστε να μπουν και σε τροχιές κοντινές προς την γη έτσι ώστε να απορροφηθούν από την ατμόσφαιρα όλο και περισσότερα αντικείμενα που μπορεί να είναι είτε δορυφόροι ε, που δεν ε, λειτουργούν πλέον, είτε απόβλητα ε, ή παράγωγα παλαιότερων συγκρούσεων. Πρόσφατα είχαμε σύγκρουση ανάμεσα σε ένα μικρό δορυφόρο της Κεντρικής Αμερικής και έναν πύραυλο της Σοβιετικής Ένωσης. της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και θα ήθελα ε, να ληφθεί υπόψη άμεσα η ευρωπαϊκή ε, βιομηχανία, διαστημική βιομηχανία είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό, είναι σε θέση να δημιουργήσει ε, δομές ε, οι οποίες θα μπορούσαν ας πούμε να είναι μικρά διαστημόπλια τα οποία θα μπορούν να κολλώνται ας πούμε κατά κάποιο τρόπο πάνω στα, στους δορυφόρους που δεν λειτουργούν πλέον και να τους οδηγούν ε, εκεί που πρέπει. Χρειάζεται πάντως ένα εξειδικευμένο κεφάλαιο, μία διεθνή συμφωνία οπωσδήποτε έτσι ώστε να καθαριστεί το ε, διάστημα. Ε, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις δορυφόρων που φτάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους αλλά δεν έχουν διαλυθεί ακόμα Λοιπόν, νομίζω ότι σε διεθνέ επίπεδο πρέπει να υπάρξει κάποια συμφωνία μεταξύ όλων των χωρών που έχουν ε, βάλει δορυφόρου ε, κατά τα διαστήματα στο, στο διάστημα. οι αρμόδιες υπηρεσίες ε, διαστήματος και αεροναυπηγικής μπορούν να βρουν περιπτώσεις σε κάποια ας πούμε μηχανήματα τα οποία θα είναι ε, μικροί δορυφόροι και οι οποίοι με έναν ε, κινητήρα μικρής ισχύω θα μπορούν ε, ιόντων ε, που, με, ε, που θα μπορούν να προσκολώνται λοιπόν όπως είπαμε σε αυτόν τον δορυφόρο έτσι ώστε να, μπορούν, να, να μπορέσει να καθαρίσει το διάστημα κάποια στιγμή από όλα αυτά τα υπτάμενα αντικείμενα. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως θα πρέπει να διέπεται από κώδικα καλής συμπεριφοράς και βελτίστων πρακτικών έτσι ώστε όταν λίγοι και ο κύκλος ζωής, ολοκληρώνει το κύκλο ζωής των δορυφόρων, να τίθενται εκτός ε, τροχιάς. Νομίζω ότι όλοι όσοι στέλνουν δορυφόρους στο διάστημα θα πρέπει να ε, ευαισθητοποιηθούν για το θέμα αυτό έτσι ώστε μετά τις δραστηριότητές τους να μένει το διάστημα όσο γίνεται πιο καθαρό. Ε, ε επίσης ένα άλλο πρόβλημα μπορεί να προκύψει από, τους... από τις ηλιακές καταιγίδε. Έχουμε δει ε, ότι υπάρχουν τέτοιες καταιγίδε πρόσφατα και έχουν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα ε, στο, στα ε, δίκτυα του ηλεκτρικού. Αυτές οι ηλιακές καταιγίδε δεν ξέρουμε ακόμα πώς λειτουργούν ακριβώς. Δηλαδή δεν ξέρουμε εάν δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα ε, σε, ε, σε μηχανισμούς που λειτουργούν ή που βρίσκονται εκτός λειτουργίας. Ε, θα, όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε γιατί η εξάρτησή μας από το διάστημα είναι υπερβολικά μεγάλη έτσι ώστε να εξακολουθούν να υπάρχουν τόσες πολλές και άγνωστες παράμετροι όσον αφορά το ίδιο το διάστημα. Ε, κάτι ανάλογο θα μπορούσε ε, να είναι και αυτό το αντικειμένο ε, των εξω, αντικειμένων που αρχίζουν και πλησιάζουν επικίνδυνα Πρόκειται για αντικείμενα τα οποία θα πρέπει να τοποθετηθούν στον χώρο με μεγάλη ακρίβεια έτσι ώστε να καθοριστεί η τροχιά τους και ε, επομένως να καθοριστεί ε, και ο κίνδυνος που αντιπροσωπεύουν για τον ε, ίδιο τον πλανήτη, για τη γη αλλά και για τους δορυφόρους. Ε, κοιτάξτε, εγώ μακρηγόρησα λίγο γιατί είναι το τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης, αλλά ε, πραγματικά ήθελα να τα πω αυτά τα πράγματα. Να πω και κάτι άλλο. Πρώτον, όσον αφορά τις επενδύσεις. Κοιτάξτε, αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, ε, ας πούμε, για το πρόγραμμα, για τον Γαλιλαίο. Ε, υπήρξε μια κοινή ε, διαδικασία ε, δημόσιου και ιδιωτικού, σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Πρέπει να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ξεκινήσει μία διαδικασία εντατική επένδυσης, επενδυτικής ε, διαδικασίας σε, αυτούς, σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει ενδεχομένως ε, να σκεφτούμε και το θέμα της ιδιωτικοποίησης ή τη σύσταση ενός ε, ταμείου ανακύκλησης που θα επιτρέπει την σωστή και διαρκή επένδυση στο διάστημα και σε όλους με αυτό σχετίζονται. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ότι όλα αυτά θα πρέπει να ε, τα δούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και να τα κοιτάξουμε και να τα μελετήσουμε υπό το πρίσμα των επενδύσεων. Γιατί στην ουσία επενδύουμε για το μέλλον μας, επενδύουμε ε, για, ε, Ευρωπές, για, συγγνώμη, για δομές οι οποίες θα είναι καθαρά ευρωπαϊκές. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ μέλλον ευρωπαϊκό χωρίς τον Γαλιλαίο, χωρίς τον Κοπέρνικο, χωρίς το, τα, στοιχεία αυτά για το μέλλον των τηλεπικοινωνιών. Πρόκειται για στοιχεία τα οποία είναι άρρηκτα συνδεμένα με το μέλλον μας. Και νομίζω ότι μπορούν αυτά τα στοιχεία να αναπτυχθούν, να πολεμήσουν την κακή συγκυρία. Ναι, μιλήσατε 9 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, λέει η Πρόεδρος, αλλά ε, σας, το, σας άφησα, όντως. Ο κύριος Σωτοζενόφσκι. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Συγγνώμη που καθυστέρησα. Άρχισα λόγω της ε, προηγούμενης ε, συνάντησης. Εγώ συμμερίζομαι όλες ε, τις, και συμφωνώ με όλες τις δραστηριότητε καινοτομία, ιδίως ό,τι αφορά το διάστημα, γιατί το διάστημα σχετίζεται και με τις νέες αναδυόμενες τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να μας βοηθήσουν και είμαι πεπισμένος ότι η έρευνα στο διάστημα είναι από τις προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί εάν η διαστημική έρευνα αποτελεί αρμοδιότητα μόνο ενός κράτους μέλους, δεν θα καταφέρει ποτέ ένα μεμονωμένο κράτος μέλος να αποκτήσει αρκετή τεχνογνωσία και να έχει το κατάλληλο προσωπικό. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ένας από του τομεί όπου βλέπουμε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Νίμπλερ. Είμαι σίγουρος ότι θα αξιοποιήσει και τις προηγούμενες εκθέσεις ως βάση για τη δική της έκθεση. Κάποια προγράμματα έχουν ήδη ξεκινήσει, για παράδειγμα ο Γαλιλαίος. Και είναι θεμελιώδη σημασία η επιτυχή έγκυβαση αυτού του προγράμματο, γιατί θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων προγραμμάτων. Και ο κόσμο θα πιστέψει ότι αυτά τα προγράμματα, παρότι μπορεί να είναι ακριβά, είναι σημαντικά. Και άλλα προγράμματα υπάρχουν που θα ανακύψουν μετά από τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Ο Γαλιλαίος θεωρώ ότι θα έχει μεγάλη επιτυχία. Ο καθηγητής Πρόντι ανέφερε κάποια προβλήματα, κρίσεις, προβλήματα ε, λόγω έλλειψης ε, εταιρικών σχέσεων συμπράξεων με τον ε, ιδιωτικό τομέα. Θεωρώ όμως ότι το πρόγραμμα Γαλιλαίος θα είναι επιτυχές. Βεβαίως θα απαιτείται και η εξέβρεση των απαραίτητων πόρων, όμως η διαστημική έρευνα είναι τομέας για τον οποίο θα πρέπει να συνεργαστούν όλα τα κράτη-μέλη για την εξέβρεση λύσεων. Χαίρομαι που η κυρία Νίμπλερ έχει αναλάβει αυτή την έκθεση, γιατί είναι ιδιαίτερα πεπειραμένη, γνωρίζει ε, πολλές λεπτομέρειες για το πρόγραμμα Γαλιλαίος Εγώ ας πούμε θεωρώ ότι πρέπει και κάποιες νέες επιχειρήσεις, οι λεγόμενες startups, ε, να συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια και με το να επενδύσουμε σε νέες τεχνολογίες θα δούμε και περαιτέρω ανάπτυξη. Η διαστημική έρευνα θα αποτελέσει κινητήριο μοχλό για αυτή την ανάπτυξη. Προσβλέπω λοιπόν σε περαιτέρω συνεργασία και ελπίζω η έκθεση να είναι επιτυχής. Χαίρομαι που μπορούμε να αποδείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να ανταγωνιστεί άλλες δυνάμεις που ασχολούνται με το διάστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τον Σάνθρο Η Κομισιόν έχει το λόγο. Εάν επιθυμεί, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε θα ήθελα να συμμεριστώ ορισμένε ιδέε με τα μέλη, να μοιραστώ ορισμένε ιδέε με τα μέλη τη Επιτροπή σα που διατρέχουν την πρόταση τη Κομισιόν. Κάποιε από αυτέ τι προτάσει αναφέρθηκαν ήδη από τα μέλη τη Επιτροπή σα. Για μένα είναι σημαντικό να τοποθετήσουμε αυτή την ανακοίνωση της Κομισιόν στο σωστό οικονομικό πλαίσιό της. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κρίση, σε μια κρίση η οποία ζητά διαρθωτικές λύσεις αλλά ζητά και παροχή κινήτρων για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα σε βιομηχανικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν είναι η πρώτη η οποία αναγνωρίζει τη σημασία που επέχει η βιομηχανία γενικά και όχι μόνο η διαστημική στη διαδικασία που θα πρέπει να μας οδηγήσει στην έξοδο του τούνελ και της κρίσης για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την οικονομική ανάκαμψη και την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Η βιομηχανική, συγγνώμη, η διαστημική βιομηχανία είναι σημαντικό τμήμα του βιομηχανικού ιστού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. <clears throat> Δίνει δουλειά σε 35 ε, χιλιάδες άτομα και τζίρο 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι ένας φυσικά τομέα σε απόλυτους αριθμούς, αλλά ένας τομέας μεγάλης και νευραλικής σημασίας στο βαθμό που δημιουργεί τεχνολογική καινοτομία η οποία μετά μπορεί να μεταλαμβατευτεί και να εφαρμοστεί σε άλλους βιομηχανικούς τομείς. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν είναι και σημαντική όπως και για τις υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες μας, όπως ανέφεραν ορισμένοι από τους ομιλητές σας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα θα πρέπει να καναγνωρίσουν τη σημασία του διαστημικού τομέα και στο βαθμό που προχωρούν οι διαπραγματεύσεις για τις πολιετήσεις δημοσιονομικές προοπτικές βλέπουμε ότι τα επόμενα 7 χρόνια θα υπάρξει σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης για τα διαστημικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Γαλιλαίος, ο Κοπέρνικος, η διαστημική έρευνα στο, στα πλαίσια του ορίζοντα 2020. Έχει κέριο χαρακτήρα η δημόσια επένδυση και χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αποτελεί το 61% του συνολικού τζίρου αυτής της βιομηχανίας. Συγχρόνως όμως, η βιομηχανία θα πρέπει να αναπτύξει και την εμπορική πτυχή της. Λειτουργεί πολύ καλά, είναι ισχυρή σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχει να αντιμετωπίσει όμως σημαντικές προκλήσεις δεδομένου ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον πλανήτη. Έχουμε τους ανταγωνιστές μας οι οποίοι και αυτοί έχουν ε, επιθετικούς στόχους. Είναι νέες δυνάμεις που αναδύονται σε παγκόσμιο επίπεδο και επομένως η Κομισιόν έχει διατυπώσει αυτή την ανακοίνωση για την διαστημική βιομηχανική πολιτική, διότι ήθελε να διακριβώσει με ποιο τρόπο θα μπορούσε να βελτιώσει το πλαίσιο στο οποίο εργάζεται αυτή η βιομηχανία για να γίνει πιο καινοτόμα και πιο ανταγωνιστική. Η κυρία Νίμπλα ήδη αναφέρθηκε στους στόχους αυτής της ανακοίνωσης της Κομισιόν, δεν θα χρειαστεί να τα επαναλάβω όλα αυτά. Προτείνει και προβλέπει τώρα η ανακοίνωση αυτή μία σειρά από δυνητικά μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με το ρυθμιστικό πλαίσιο, το κανονιστικό πλαίσιο καλύτερα, για να λειτουργήσει καλύτερα η διαστημική βιομηχανία, προβλέπει την, την υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης, μορφές χρηματοδότησης <clears throat> και υποστήριξης πέραν των καθαρά προγραμματικών, μια υποστήριξη από την θεσμική αγορά, επίσης και υποστήριξη στα θέματα των εκτοξευτών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί εδώ έρχομαι σε αυτά που είπε ο κ. Πρόδη. Το θέμα της προστασίας των διαστημικών υποδομών. Η Κομισιόν έχει παρουσιάσει μια πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτή γιατί γνωρίζει <clears throat> την ανάγκη να υπάρξει προστασία αυτών των υποδομών στο διάστημα και η Επιτροπή σας θα έχει την ευκαιρία να αντιμετωπίσει λίγαν προσεχώς με την πρωτοβουλία αυτή που προέρχεται από την Κομισιόν και έχει σαν στόχο να δημιουργηθεί ένα σύστημα έγκαιρες προειδοποίησεις για συγκρούσεις στο διάστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, τα προγράμματα έρευνας στο διάστημα περιλαμβάνουν σχέδια τα οποία προωθούνται και τα οποία έχουν σαν στόχο το να καθαρίσουν τα απόβλητα, τα διαστημικά που κυκλοφορούν, δύο σε χαμηλές τροχές. Ελπίζουμε λοιπόν ε, αν μπορώ να το πω αυτό, την θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, όπως είπε και η κυρία Νίμπλερ, να δούμε ποιες είναι οι απόψεις των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τις προτάσεις που περιέχονται στην πρόταση της Κομισιόν. Ίσως κάποιες αυτές τις προτάσεις είναι πιο ενδιαφέρουσες από άλλες. Γι' αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και η δική σας γνώμη. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ την Κομισιόν. Τον ε, λόγο θα έχει η συνάδελφος Νίμπλερ για να κάνει τι τελικέ της παρατηρήσει. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους οι οποίοι έλαβαν το λόγο και έδωσαν προτάσεις και ιδέες για την έκθεση και επίσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά που ανέφερα. Νομίζω ότι σε πρώτη ανταλλαγή απόψεων γίνεται πάρα πολύ σημαντικό πόσο μεγάλη στρατηγική σημασία που έχει διαστημική πολιτική για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και ποια είναι η σημασία που πρέπει να αποκτήσει, ακόμα και ένας μικρός τομέας ο οποίος δεν έχει πάρα πολλούς εργαζόμενους. Νομίζω ότι από στρατηγική έποψη μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο για όλη τη βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ακριβώς και το θέμα του πώς πρέπει να εξασφαλιστούν οι επενδύσεις στον τομέα αυτό. Και όπως είπε και ο κύριος Πρόντι, ακριβώς λόγω της κρίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε την διαστημική βιομηχανία. Είδαμε ότι το σύστημα των εταιρικών σχέσεων δημόσιου ιδιωτικού τομέα δεν λειτουργήσε πάρα πολύ καλά στην περίπτωση του Γαλιλαίου. Πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν τα απαραίτητα κίνητρα για να τονώσουμε τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και να βελτιώσουμε την κατάσταση σε σχέση με αυτά που είδαμε στον Γαλιλαίο. Το θέμα της συλλογής των απορριμμάτων στο διάστημα είναι ένα δύσκολο θέμα, αναφέρθηκε από όλους σας και αυτό είναι ένα ζήτημα ε, το τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη στον τομέα αυτό. Εμείς λοιπόν πρέπει καταρχήν να έχουμε ένα σύστημα επαγρύπνησης για τα απορρίμματα τα οποία κινούνται στο διάστημα για λόγους ασφαλείας των υποδομών των διαστημικών και νομίζω ότι και αυτό αναφέρεται στην ε, ε ανακοίνωση της Κομισιόν αλλά ίσως υπερβολικά σύντομα. Νομίζω ότι με τη βοήθεια των συναδέλφων πρέπει να ενισχύσουμε αυτές τις προτάσεις και να καταθέσουμε θέσεις και προτάσεις για το ζήτημα αυτό που είναι ένα ζήτημα το οποίο αξίζει περισσότερη ε, προσπάθεια από την πλευρά. Όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, είναι σημαντικό να έχουμε αυτό το σύστημα που αποτρέπει τις συγκρούσεις και φυσικά θα πρέπει να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις λεπτομέρειες στο ζήτημα αυτό. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους. Όλοι μας παρακολουθούμε το σχέδιο Γαλιλαίος εδώ και πολύ καιρό με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον και τα άλλα προγράμματα όπως ο Κοπέρνικος και αυτά είναι θέματα τα οποία εμπλέκονται και στον ορίζοντα 2020 τα οποία συζητούνται και στον ε, τριμερή διάλογο Νομίζω λοιπόν ότι μπορώ προς το παρόν να σας ευχαριστήσω για, την, για τις απόψεις που έχετε διατυπώσει και χαίρομαι γιατί αυτό το θέμα, αυτά τα θέματα παρακολουθούνται από πολλούς συναδέλφους εδώ και πολύ και χρονικό διάστημα που εξέφρασαν ήδη και την άποψή του. Είμαστε λίγοι αλλά θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και να εκφράσω, εκφράσω και το σεβασμό μου για ένα από τους συναδέλφους μας ο οποίος έχει βρεθεί ήδη στο διάστημα και επίσης και στον κύριο Πρόντι ο οποίος ασχολείται με το θέμα αυτό τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί τόσο στενά για, αυτήν, για προηγούμενες εκθέσεις και ελπίζω και σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ελπίζω λοιπόν όπως είπατε κυρία Πρόντι, να μπορέσουμε να κλείσουμε αυτό το θέμα εφέτος. Ευχαριστούμε πολύ την ε, συνάδελφο Νίμπλερ. Ολοκληρώσαμε τις ε, εργασίες μας. Στις 5.30 ε, θα λάβει χώρα εδώ η συνεδρίαση των συντονιστών. Να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι 9 το πρωί αύριο θα ξαναρχίσει η πρωινή μας συνεδρίαση με ψηφοφορίες. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.